Hello, I'm uh, a... Γεια σας, κυρίες μου και κύριοι, κύριε τουλάχιστον. Παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε αργήσει επειδή αργήσαμε λίγο στο κύριο πάνελ αλλά ο χρόνος πιέζει γι' αυτό θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αγαπητοί ευρωβουλευτές, δεν ξέρω πόσοι υπάρχουν, κάποιοι θα είναι, αγαπητοί βουλευτές, συνάδελφοι και φίλοι, με χάρα σας καλωσορίζω στο εργαστήριο το οποίο είναι αφιερωμένο στην ε, χάραξη πολιτικής που λαμβάνει υπόψη την διάσταση του φίλου και βρίσκεται στην καρδιά της ε, ανάπτυξης ε, με συμπερίληψη. Λοιπόν, να σας πω τι θα γίνει, πώς θα μιλήσουμε. Θέλω να δώσετε στους κλητήρες τις κάρτες σας για να μιλήσετε που θα γράφουν το όνομά σας και το κοινοβούλιο από το οποίο είστε. Μπορείτε να τις δώσετε τα επόμενα 15 λεπτά, πρέπει να είναι μπροστά σας ε, πάνω στα έδρανα. και σε 15 λεπτά θα κλείσει ο κατάλογος των ομιλητών. Να ξεκινήσουμε λοιπόν αμέσως με την ομιλήτριά μας σήμερα, την κυρία Τατιάνα Τέπλοβα από τον ΩΣΑ, η οποία είναι υποδιευθύντρια για τις ε, αξιολογήσεις ε, της ε, διακυβέρνησης και της, ε, του διαχωρισμού αρμοδιοτήτων και βεβαίω αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνη για την ισότητα των φύλων στη δημόσια ζωή, στον ΩΣΑ και προωθεί διεθνείς ε, προδιαγραφές για την σχετική πολιτική, για την επέκταση των δεδομένων με ανάλυση αναφύλο για την προώθηση του διαλόγου και για την ενίσχυση της θεσμικής και νομικής δυνατότητας ε, ισότητας ε, των φίλων. Ε, πολύ σοβαρή η δουλειά σας ε, και πολλά τα καθήκοντά σας. Λοιπόν, έχετε τον λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι και αγαπητοί προσκεκλημένοι, είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για εμάς στον ΩΣΑ το ότι οργανώνουμε αυτό το εργαστήριο μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Διεθνή ημέρα των γυναικών και θα εστιάσουμε όπως είπαμε στο πως ε, λαμβάνεται υπόψη η διάσταση των φύλων ε, στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης ε, και της ανάπτυξης με συμπερίληψη. Θα ξεκινήσω λοιπόν μιλώντας για το κενό, τον, το χάσμα των φύλων και τα εργαλεία τα οποία έχουμε για τη χάραξη τέτοιας πολιτικής και τον ρόλο που μπορούν να παίξουν τα κοινοβούλια σε αυτήν. Λοιπόν, συνολικά, όπως ε, ακούσαμε και νωρίτερα, φαίνεται ότι υπάρχει κάποια πρόοδος ε, προς την ισότητα, αλλά υπάρχουν ακόμα κάποια κένα. Εάν δούμε τις χώρες μέλη του ΩΣΑ, που είναι 35 αυτή τη στιγμή, λίγο περισσότερες από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν την βία με βάση το φύλλο, το χάσμα των αμοιβών. Επίση, το πώς θα διαμοιράζεται η απλήρωτη εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών και η πρόσβαση σε θέσεις ε, ηγεσία και όπως αναφέρθηκε και από άλλους ε, διακεκριμένους ομιλητές η βία βεβαίως παραμένει η πρώτη προτεραιότητα, αλλά τα δεδομένα είναι λίγα. Ξέρουμε ότι μία στι τρει γυναίκες ανά την υφήλιο έχει, υφίσταται κάποια μορφή βία, είτε σεξουαλική είτε σωματική, είτε από τον σύντροφό τη είτε από άλλους. Και Βλέπουμε και βεβαίως και άλλες ψαλίδες όπως την εκπροσώπηση των γυναικών στο Κοινοβούλιο όπου ε, υπάρχει κάποια πρόοδος αλλά η ψαλίδα παραμένει. Οπότε εάν δούμε όλα τα μέλη του ΩΣΑ βλέπουμε ότι σε σύγκριση με το 2002 το 2016 είχαμε μία αύξηση, δεν θα έλεγα σημαντική αλλά τέλος πάντων είναι μία βελτίωση. Σήμερα δηλαδή είμαστε στο 28% 100, κάτω από το 30% αλλά είναι μια βελτίωση ε, κατά 20% σε σχέση με το 2002. Και αυτό είναι βεβαίως ε, προβληματικό όταν μιλάμε για τα κοινοβούλια γιατί τα δικά σας ε, ακριβώς αυτά τα θεσμικά όργανα νομοθετούν. Χαράζουν δηλαδή τους κανόνες ε, και τις ε, διαδικασίες ε, πρόσβασης σε ιδιωτικούς και δημόσιους πόρους ε, και εκπροσωπούν και την κοινωνία που υπηρετούν. Αν πάμε λοιπόν στην επόμενη διαφάνεια, η κατάσταση εκπροσώπησης των γυναικών μεταξύ των προέδρων των κοινοβουλίων είναι ακόμη πιο ανησυχητική. Γύρω στο 21% των προέδρων κοινοβουλίων ε, είναι γυναίκες και η Ολλανδία είναι η μόνη χώρα του ΩΣΑ όπου η πρόεδρος ε, της Άνω και της Κατοβουλής είναι γυναίκες. Μια παρόμοια κατάσταση βλέπουμε και στη δικαιοσύνη. Αν δούμε τα δύο διαφάνειες πίσω Αν δούμε λοιπόν τους ανώτατους δικαστικούς, υπάρχουν ε, αρκετές γυναίκες, 54% ε, δικαστίνες ε, στα κατώτερα δικαστήρια, οπότε υπάρχει υπερεκπροσώπηση θα λέγαμε στις κατώτερες βαθμίδες, αλλά εάν δούμε τα ανώτατα δικαστήρια, βλέπουμε ότι οι γυναίκες έχουν μόνο 33% 0,6% των θέσεων στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας του ΩΣΑ και κατά μέσο όρο όταν μιλάμε για τις προεδρίες των δικαστηρίων έχουμε μια παρόμοια εικόνα. Στα κατώτερα δικαστήρια οι γυναίκες είναι στο 45,9 σχεδόν 50% δηλαδή προέδρων δικαστηρίων στα εφετεία, ας πούμε, χοντρικά, είναι γύρω στο 1 τρίτο οι πρόεδροι γυναίκες και όταν μιλάμε για τα ανώτατα δικαστήρια μιλάμε για 18,6%. Όσον αφορά τώρα τον δημόσιο τομέα, η εικόνα είναι παρόμοια. Εκπροσωπούνται πολλοί γυναίκες στο δημόσιο τομέα, αλλά όταν μιλάμε για τις θέσεις της ε, Διοίκηση εξακολουθεί να υπάρχει χάσμα και είναι γύρω στο 1 τρίτο των ε, θέσεων ε, των υψηλόβαθμων. Και στην ευρύτερη οικονομία όταν μιλάμε για την συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας βλέπουμε κάποιες βελτιώσεις κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας αλλά το χάσμα Τη συμμετοχή ανδρών και γυναικών ε, παραμένει γύρω στο 8,5% και Βεβαίω ε, αυτό το οποίο δεν έχουν η δυσκολία στις γυναίκες να ανέλθουν στα ανώτατα αξιώματα είναι ακόμη μεγαλύτερη σε σχέση με την δημόσια ζωή. Αν δούμε παραδείγματος χάρη τις εισηγμένες εταιρείε ε, και τις κορυφαίες θέσεις εκεί είναι ακόμα πολύ απόμακρος ο στόχος. Το 2016 στον ΟΣΑ 20% των μελών διοικητικών συμβουλίων είναι γυναίκες και αν δούμε τους διευθύνοντες συμβούλους μιλάμε για 4,8% που είναι γυναίκες. Αλλά και τα δύο αυτά νούμερα είναι σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2013 όταν ήταν 16,4 των μελών διοικητικών συμβουλίων και 2,4 των ε, συμβούλων. Τώρα η διαφορά στους μισθούς, το είπανε και προηγούμενοι ομιλητές. Είναι μεγάλη προτεραιότητα για τις χώρες μας και είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει η κατάσταση εδώ. Σε όλες τις χώρες του ΩΣΑ βλέπουμε ότι είναι επίμονο γύρω στο 15% αυτή η διαφορά στις αμοιβέ. Βελτιώθηκε κάπως κατάσταση στην ε, Χιλή, τη Λουθουανία, το Μεξικό και την Πορτογαλία. Αλλά στην Σλοβενία αυξήθηκε το χάσμα των μισθών, η διαφορά των μισθών. Αυτά τα χάσματα ε, με βάση το φύλλο θίγουν τους πάντες, και τις άνδρες και τις γυναίκες, και έχουν και ισχυρό αντίκτυπο στην κοινωνία. Και μπορούμε να το δούμε από πολλές διαφορετικές απόψεις. Από οικονομική πλευρά το χάσμα της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, αν μειωθεί στο μισό, αν πάει στο 20-25% τότε θεωρούμε ότι το ΑΕΠ σε όλες τις χώρες του ΩΣΑ κατά μέσο όρο θα αυξηθεί κατά 12%. Σαφές λοιπόν οικονομικό επιχείρημα για να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Και τι μας δείχνει αυτή η διαφάνεια επίσης. Ότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ της συμμετοχής των γυναικών σε πιο ανώτερες θέσεις, σε διοικητικά συμβούλια και εδώ στο επίπεδο, εδώ είναι κυρίως για τα Υπουργεία αυτό αυξάνει την εμπιστοσύνη της κοινή γνώμης στους δημόσιους θεσμούς. Και επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ του αριθμού γυναικών μεταξύ των βουλευτών και της μείωσης της ε, ανισότητας. Βέβαια, οι ακριβείς λόγοι για αυτό το συσχετισμό ε, είναι δύσκολο να ανοιχνευθούν και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην ερμηνεία μας. Αλλά εξετάζοντας την κατάσταση σε μεμονωμένες χώρες, διαπιστώνουμε ότι πολύ συχνά οι γυναίκες νομοθέτες αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη μείωση του χάσματος με βάση το φύλλο και αυτά βεβαίως ωφελούν ε, ευρύτερα την κοινωνία. Για παράδειγμα, στην πρόσφατη εξέταση της κατάστασης ε, στο Μεξικό για την κατάσταση με βάση το φύλλο στο Μεξικό λοιπόν είδαμε ότι 85% των νομοθετημάτων που προσπαθούσαν να προωθήσουν την ισότητα προτάθηκαν από γυναίκες βουλευτές. Είναι δύσκολο να βρούμε τη σχέση αιτίου αποτελέσματος, αλλά βλέπουμε σημαντικό αντίκτυπο ανάμεσα σε διάφορα φαινόμενα. Άρα τι μπορούμε να κάνουμε. στις χώρες του ΟΣΑ και μάλλον όχι, στον οργανισμό ΟΣΑ και ιδιαίτερα στην διεύθυνση για τη διακυβέρνηση διαπιστώνουμε ότι η πολιτική με βάση την ευαισθησία για το φύλλο παίζει μεγάλο ρόλο γενικότερα. Μέσω της απόδοσης πόρων, διαφόρων πολιτικών, διαφόρων νόμων μπορούμε να προωθήσουμε ή να εμποδίσουμε την ισότητα και μπορούμε λοιπόν να έχουμε θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα. Και το επιχείρημά μας είναι ότι πρέπει τα θέματα φύλου να είναι στην καρδιά όλων των ενεργειών των κυβερνήσεων, όλων των αποτελεσμάτων των νομοθετημάτων και των πολιτικών και στη διαδικασία λήψης όλων των αποφάσεων. Έχουμε εδώ μάλιστα και ένα έντυπο το οποίο εκδόθηκε πριν από δύο χρόνια και που εξακολουθεί να είναι επίκαιρο, που δίνει σε βάθος ανάλυση των δεδομένων. Και εδώ έχουμε και τις νέες συστάσεις, που περιγράφουν μια σειρά από μέσων και εργαλείων που έχουμε και έναντι των κοινοβουλίων για να προωθηθεί η διαμόρφωση πολιτικής που λαμβάνει υπόψη το φύλλο. Και μπορούμε να διαχωρίσουμε τρεις κύριους άξονες. Πρώτον, μέτρα για να κλείσει το χάσμα στην εκπροσώπηση στους δημόσιους θεσμούς μεταξύ των φίλων, ιδιαίτερα μεταξύ των ε, ε, ε, ατόμων που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Επανέρχομαι σε αυτό το θέμα ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις. Το δεύτερο είναι να υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που να διαχωρίζουν αναφύλο για να βοηθήσουν ακριβώς αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις να κατανοήσουν την επίπτωση των νέων νομοθετημάτων, των νέων πολιτικών, αλλά και τα αποτελέσματα των ήδη ε, ισχυουσών πολιτικών. Και τρίτον, αποτελεσματικοί θεσμικοί μηχανισμοί και πλαίσια. Και αυτά μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο. Εσείς, ως κοινοβουλευτικοί, βεβαίως μέσω νομοθετημάτων, μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου και μέσω του ρόλου προτύπων που παίζετε, μπορείτε να έχετε μια σημαντική επίπτωση. Τώρα, οι συστάσεις μας αυτές αναφέρουν διάφορες εναλλακτικέ ε, δυνατότητες για να τις εξετάσετε ανάλογα με τη χώρα για τις χώρες που ε, προσπαθούν να μειώσουν αυτό το χάσμα εκπροσώπησης ε, στα δημόσια όργανα. Τώρα δεν θα τα αναφέρω αναλυτικά, στη διάθεσή σας για να τα συζητήσουμε. Να τονίσω όμως ίσως ορισμένα θέματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να, ασχολούμε, να ασχοληθούμε και με την πλευρά της ε, προσφοράς, δηλαδή να αυξηθεί η ορατότητα των γυναικών. Είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες που έχουν προσόντα, που έχουν δεξιότητες, να έχουν τη θέληση να καταλάβουν ηγετικές θέσεις σε δημόσιους ε, οργανισμούς και φορείς. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει πολύ σημαντική δουλειά και το Κοινοβούλιο συγκεκριμένα για να προωθήσει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου. Θέλω να τονίσω τα εξή σημεία. Πρώτον, η, αυτά τα προγράμματα ισορροπίας μεταξύ ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου πρέπει να αφορούν και τις ε, ηγετικέ θέσεις. Τα ευέλικτα, τα ελαστικά ωράρια, οι γονικές άδειες, οι άδειες μητρότητας, όλα αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα και για αυτούς που είναι στο υψηλότερο επίπεδο, που λαμβάνουν τις ε, κύριες αποφάσεις. Αυτό αναφέρθηκε και ως πόρισμα της έρευνάς μας. Οι γυναίκες πολύ δεν έχουν ε, ούτε καν ε, τη διάθεση να καταλάβουν ηγετικές θέσεις γιατί θεωρούν ότι θα έχουν πρόβλημα στην ε, προσωπική τους ζωή. Δεύτερο θέμα. Πρέπει να ενθαρρύνουμε και τους άνδρες να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες. Δεν είναι δηλαδή αποκλειστικά οι γυναίκες που θα πρέπει να ωφελούνται από αυτές τις δυνατότητες. Γιατί αυτό τελικά μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις κατά των ανδρών. Και τρίτον, Πρέπει να θαρρύνουμε και τους άνδρες και τις γυναίκες να μοιράζονται καλύτερα την απλήρωτη εργασία και την ευθύνη της ανατροφής των παιδιών. Γιατί βεβαίως ε, ε, αυτά που προτείνουμε εμείς είναι επίσημες αλλαγές μέσω νομοθετημάτων και κανόνων. Αλλά αν δεν υπάρχει καλύτερη κατανομή της, ε, των εργασιών στο σπίτι και για την ανατροφή των παιδιών, είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθούν όλα αυτά. Τώρα ακόμη πιο σύντομα θα αναφερθώ στα επόμενα θέματα για τις χώρες και για τους πολιτικούς ευθύνοντες και πώς μπορούν να προωθήσουν μια πολιτική και όλες τις πολιτικές με πιο πολλές ευαισθησίες ό,τι αφορά τη διάσταση του φύλου. Εδώ να τονίσω τις ε, μελέτες αντικτύπου ό,τι αφορά το φύλο. Ουσιαστικά δηλαδή τα αναλυτικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται για να γίνει αντιληπτό ο αντικτύπο των πολιτικών, των ε, των επιδοτήσεων στη θέμα τη διαστασία του φύλου. Τι βλέπουμε λοιπόν στη διαφάνεια. 25, 25 χώρες του ΩΣΑ έχουν εγκρίνει υποχρεωτική εφαρμογή των ε, θεμάτων του φύλου στους κανονισμούς και στην νομοθεσία. Θα μας ενδιαφέρει λοιπόν να δούμε τι γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα εθνικά σας κοινοβούλια. Δηλαδή, πώς οι νομοθέτες χρησιμοποιούν και αξιοποιούν τα εργαλεία αυτά τα οποία την ανάλυση. Τώρα, να δούμε το θέμα της χρηματοδότησης σε ό,τι αφορά τη διάσταση του φύλου. Εδώ θεωρώ ότι πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο έχει λάβει κάποια προβολή, μεν, αλλά ακόμα δεν αξιοποιείται πλήρως και ουσιαστικά έχει να κάνει με το gender mainstreaming, ε, δηλαδή με την προσαρμογή στη διάσταση του φύλου σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό και τη χρηματοδότηση. Σε διάφορα επίπεδα της, ε, του προγραμματισμού για τη χρηματοδότηση. Γιατί λοιπόν είναι σημαντικό αυτό. Γιατί βλέπουμε ότι πολλές από τις διαφορές και τις ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών προκύπτουν ακόμα, ακόμα και στις βασικές θεμελιώδεις πολιτικές και χρηματοδοτήσεις οι οποίες συντηρητούνται επί χρόνια. Και αυτό λοιπόν βοηθά πάλι με τη σειρά του να κατανοήσουν οι χώρες και να επιλύσουν κάποια από τα προβλήματα που προκύπτουν σε ό,τι αφορά το χάσμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση, την ίση ανάλογα με τα φύλλα, βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια πρόοδος. Περιορισμένη. Αυτό το gender budgeting λοιπόν έχει εισαχθεί σε Αρκετές χώρες του ΩΣΑ και κάποιες άλλες το σκέφτονται ακόμα, αλλά το θέμα είναι ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία θα μας επιτρέψουν να καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται και ποιος είναι ο αντικτύπος. Τέλος. Τα θεσμικά όργανα παίζουν σημαντικό ρόλο για να αντιληφθούμε ποια ακριβώς είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη διάθεση του φύλου. προκειμένου τελικά να υπάρχει και σωστή εκπλήρωση των δεσμεύσεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Επιτροπή ε, για το φύλλο που εφαρμόζουν και κανόνες σε ό,τι αφορά τη σύνθεση τους, ε, σε ό,τι αφορά τα φύλλα, γίνονται όλο και πιο πολύ γνωστές. Και υπάρχουν και, άλλες ε, και άλλοι τρόποι για να προωθηθεί η διάσταση αυτή και με χαρά θα το συζητήσουμε. Τι μπορεί να κάνει τώρα όσα για να υποστηρίξει τις χώρες, για να υποστηρίξει όλους εσάς για να καλύψουμε αυτό το χάσμα μεταξύ των φίλων. Ανέφερα μια σύσταση η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο για την ισότητα των φίλων στη δημόσια ζωή. Έχουμε και μια σημαντική σύσταση για την ισότητα των φίλων στην απασχόληση, στην εκπαίδευση και στο επιχειρήν, στον επιχειρηματικό κόσμο. Για να εντοπιστούν οι διάφορες συναλλακτικές λύσεις που έχουν στα χέρια τους τα κράτη για να καλύψουν ακριβώς το χάσμα αυτό. Οι συνάδελφοί μου λοιπόν από τον ΩΣΑ είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή και την υλοποίηση των συστάσεων αυτών. Έχουμε επίσης πιο στοχευμένες αναθεωρήσεις και αξιολογήσεις σε ό,τι αφορά τη διάσταση του φύλου για κάθε χώρα, συλλογή δεδομένων. Μπορεί να έχετε λάβει κι εσείς ε, την ανάλυση, την έρευνα του ΩΣΑ για τις πρακτικές που είναι σχετικές με τη διάσταση του φύλου. Γίνεται τέτοια συλλογή στοιχείων και στη δημοσιοδίκηση και στο δικαστικό σώμα και βλέπουμε πόσο αποτελεσματικά είναι τα θεσμικά πλαίσια και φυσικά με χαρά θα υποστηρίξουμε την υλοποίηση όλων αυτών των συστάσεων. λέμε να αναπτύξουμε μια εργαλειοθήκη μάλιστα. Με σκοπό να εντοπιστούν οι βέλτιστες πρακτικές και να κοινοποιηθούν σε όλους benchmarks, ορόσημα, δείκτες, προκειμένου όλοι μαζί να βοηθήσουμε για να καλυφθεί το χάσμα αυτό στην Ισλανδία. Κάτι σημαντικό να αναφέρεται το Μάιο του φετινού έτου. Θα εξεταστούν οι βέλτιστες πρακτικέ και οι προκλήσει που αφορούν τη χρηματοδότηση ανάλογα με τη διάσταση του φύλου και την ένταξη τη διάσταση του φύλου σε όλε τι πολιτικέ εγκάρσια. Ευχαριστούμε λοιπόν την κυβέρνηση τη Ισλανδία για την προσπάθεια αυτή. Θα είναι σημαντική η εκδήλωση αυτή και φυσικά εσείς ως βουλευτές έχετε ιδιαίτερο ρόλο να διδραματίσετε στη συζήτηση αυτή και με χαρά θα σας υποδεχτούμε και στο Παρίσι την Παρασκευή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και με χαρά θα, ευχαριστώ, θα απαντήσουμε τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μας δώσατε πραγματικά πολύ σημαντικές πληροφορίες και όπως πάντα είμαι εντυπωσιασμένη από τις στατιστικές ικανότητες του ΩΣΑ. Επτά ομιλητές έχουμε. Και μας πιέζει και ο χρόνος. Οκτώ, οκτώ ομιλητές. Οκτώ άτομα έχουν ζητήσει το λόγο. Θα σας παρακαλούσα να μην ξεπεράσετε το 1,5 λεπτό. Για να δώσουμε και στο τέλος το λόγο πάλι στην κυρία Τέπλοβα για να απαντήσει και στα σχόλιά σας. Μάρθα Μάτρου. Έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η πολιτική της ισότητας ε, ξεκίνησε με τον διαφωτισμό όταν ο Ρουσό το έργο του Ελοΐζ ζήτησε την ίση μεταχείριση των γυναικών. Κοιτάξτε, εμείς μιλάμε για ίση μεταχείριση με τους άντρες, αλλά στο συντηρητικό μυαλό της ε, Ουγγαρίας. Δεν υπάρχει κάποια σύγκρουση εδώ πέρα. Είναι εταίροι άνδρες και γυναίκες ε, και η Ουγγρική κυβέρνηση εγγυάται τις ίσες ευκαιρίες ανδρών και γυναικών ε, και στηρίζει την γυναίκα και συνταγματικά. Η κυριότερη απειλή σήμερα είναι ότι με την μετανάστευση ε, δικαιολογούμε κάποιου από του ε, νέου ερχόμενου που παραβιάζουν τι ίσε ευκαιρίε και δεν αγκαλιάζουν αυτέ τι αξίε. Πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι όσοι έρχονται σε μια κοινωνία με ίσε ευκαιρίε πρέπει να το αποδέχονται αυτό. Η Ουγγαρία είναι μια νησίδα ειρήνη ε, μέσα σε έναν ταραγμένο ωκεανό. Και επίσης έχουμε και ένα κοινωνικό μοντέλο που βασίζεται στην οικογένεια και τις ίσες ευκαιρίες ε, σε τα κοινωνικά στρώματα και βεβαίως πρέπει να υπάρχει και πολιτική στήριξη, δέσμευση της κυβέρνησης, αλλά και συζητήσεις για να πλησιάσουμε τον στόχο αυτόν. Γι' αυτό χρειαζόμαστε προσπάθειες, ε, καλή βούληση, σαφήνεια και βεβαίω προσήλωση στους στόχους μας όπως δείχνει και αυτή η συνάντηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στην κυρία Ηλίνα Χουίστη από την Γεωργία. Ε, εγώ δεν ζήτησα το λόγο, αλλά εντάξει. Σύντομα λοιπόν είμαι από το Κοινοβούλιο της Γεωργίας έχουμε και ένα Συμβούλιο Ισότητας ε, στην χώρα που συζητά το θέμα της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και ο αριθμός των γυναικών ε, βουλευτών έχει αυξηθεί λίγο αλλά είναι ακόμα πολύ χαμηλός αλλά αντιλαμβανόμαστε επίσης ε, πλήρως ότι η συμμετοχή των γυναικών δεν θα αυξηθεί εάν δεν υπάρξει οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών. Γι' αυτό πρέπει να προωθήσουμε προγράμματα που θα βοηθήσουν τις γυναίκες να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητες και έτσι να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να ξεκινήσουν μια πιο ενεργή οικονομική και πολιτική ζωή. Είναι λοιπόν ένα περίπλοκο ζήτημα και προσπαθούμε να δούμε και το θέμα των ποσοστώσεων. Οι ποσοστώσεις είναι ένα μέτρο αύξησης της συμμετοχής. Αντιλαμβανόμαστε ότι βεβαίως μακροπρόθεσμα έχει σημασία να έχουμε, όπως σας είπα, μια οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών. Το ερώτημα λοιπόν που θα ήθελα να θέσω είναι ποιες είναι οι εμπειρίες άλλων χωρών στην Ευρώπη ως προς αυτό και πώς μπορούμε να προωθήσουμε το θέμα των ποσοστώσεων σε όσους δεν έχουν πίστη να στηρίξουν αυτό το προσωρινό μέσο αύξησης της ε, συμμετοχής των γυναικών. Σας ευχαριστώ. Ε, και για μας εδώ είναι πολύ βασικό θέμα και εντό του κομματός μου ως φιλελεύθερη εγώ βεβαίως είμαι υπέρ των ποσοστώσεων. Γιατί θα μπορούσα να πω ότι η φεμινιστική μου καρδιά είναι υπέρ των ποσοστώσεων, αλλά είναι μάχη. Και τώρα η κυρία Μαριέλα Αριστίδο από την Κύπρο. Είναι γεγονός αναφυσβήτητο ότι τα ζητήματα που αφορούν την ισότητα των γυναικών και των αντρών σε ολόκληρο τον κόσμο ποικίλουν και διαφοροποιούνται από ήπειρο σε ήπειρο, από χώρα σε χώρα, από κοινωνία σε κοινωνία Όσον αφορά την Κύπρο, παρά την αυξανόμενη ενεργό συμμετοχή γυναικών στην πολιτική και δημόσια ζωή, οι γυναίκε εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε σημαντικέ θέσει λήψη αποφάσεων. Επί του παρόντο, οι Κύπριες γυναίκε επιβαρύνονται περισσότερο από την οικονομική κρίση, διότι αναλαμβάνουν δυσανάλογο μερίδιο του νοικοκυριού, τη φροντίδα των παιδιών και των οικογενειακών ευθυνών. Συναφώ είναι επίγουσα ανάγκη να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειε για την καλύτερη συμφιλίωση τη επαγγελματική και οικογενειακή οικογενειακής ζωής μέσω της παροχή πρόσιτων και ποιοτικών υπηρεσιών οι οποίες θα είναι φιλικές προς την οικογένεια και την παιδική μέρημνα. Επιπλέον είναι υψίστη σημασία η ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, της ανάπτυξη, της υλοποίησης και της αξιολόγηση των δημοσίων πολιτικών και του προπολογισμού, αλλά και να ενισχυθούν οι μηχανισμοί λογοδοσίας και εποπτείας στον τομέα τη ισότητα των φύλων. Εν κατακλείδη, είναι απαραίτητο να επενδυθούν επαρκείς ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι και να κινητοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί σε όλα τα επίπεδα με συνέργειες και συνεργασίες. Είμαι βέβαιη ότι υπάρχει απαραίτητη αποφασιστικότητα και πολιτική δέσμευση για τον σκοπό αυτό. Σας ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε. Η επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Σιμώνα Πέτρη από τη Σλοβακία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ εκπρόσωπο το Κοινοβούλιο της Σλοβακίας Δύο πρακτικές ερωτήσεις έχω να θέσω. Η πρώτη. Μίλησατε για την ε, εργασία που δεν αποζημιώνεται, χωρίς μισθό, για παράδειγμα στο σπίτι, η φροντίδα των παιδιών και αυτό στη Σλοβακία που θεωρώ ότι δεν φύγεται ε, επαρκώς, ε, δεν προβάλλεται επαρκώς και αποτελεί αυτό ένα από τους βασικούς λόγους που δεν υπάρχει ισότητα στην κοινωνία μας. Ρωτώ λοιπόν, τι συγκεκριμένα βήματα, τι συστάσεις μπορείτε να μας κάνετε, τι βέλτιστες πρακτικές μπορείτε να μας αναφέρετε από άλλες χώρες για το θέμα ακριβώς αυτό. Για να υπάρχει καλύτερος καταμερισμός και διανομή, αν θέλετε, της απλήρωτης εργασίας. Και δεύτερο θέμα, ίσως και πιο πρακτικό ακόμα ζήτημα, κοιτάξτε την παρουσίασή σας το θέμα της συλλογή δεδομένων και εφαρμογής και ότι ο ΣΑΠ προωθεί τις βέλτιστες πρακτικές. Αυτές οι βέλτιστες πρακτικές πού βρίσκονται όμως, σε κάποιο φυλάδιο και αν υπάρχει κάποιο τέτοιο φυλάδιο όντω, πώς μπορώ να το βρω και από πού. Ευχαριστώ πολύ. Για το θέμα της απλήρωτης εργασίας θεωρώ ότι αποτελεί τις μεγαλύτερες ε, προκλήσεις και όταν έγραψα αυτό το διδακτορικό μου πριν από κάποια χρόνια το ένα τέταρτο της δουλειάς και της εργασίας όλο τον κόσμο πληρώνονται και τρία τέταρτα δεν πληρώνονται. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Η κυρία Ναπίκη από την Τινησία έχει τώρα το λόγο. Thank you, Mrs. Ευχαριστώ. Είμαι από το Κοινοβούλιο της Τινησίας. Είμαι στην Επιτροπή Δικαιωμάτων και Ελευθεριών και στην Επιτροπή Γυναικών. Σας ευχαριστώ για αυτά που μας είπατε. Επιβεβαιώνω ότι χρειαζόμαστε θαραλέους νομοθέτες. Και αυτό κάναμε στην Τινησία όταν ζητήσαμε ισότητα σε όλες, σε εκπροσώπηση δηλαδή, σε όλες τις ε, εκλεγμένες, ε, σε όλα τα εκλεγμένα σώματα. Όμως, η πραγματική πρόκληση είναι η παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, στα σώματα που λαμβάνουν αποφάσεις. Γι' αυτό πιέζουμε την κυβέρνηση να ορίσει μια επιτροπή που να εξετάζει την ισότητα των φίλων. και ελπίζω ότι θα το επιτύχουμε. Το άλλο θέμα είναι βεβαίως ε, η διαφορά στις αμοιβέ. Στις χώρες μου, στη χώρα μου συγγνώμη, αφορά κυρίως τις χαμηλόμιστες ε, γυναίκες που εργάζονται στην Γεωργία για παράδειγμα και οι οποίες δεν είναι συνδικαλισμένε. Είναι λοιπόν ε, πολύ δύσκολο να επιτευχθεί πρόοδο. Αρκεί μόνο η νομοθεσία δεν νομίζω. Πώς θα μπορέσουμε να απευθυνθούμε σε αυτές τις γυναίκες. Πώς θα μπορέσουμε να τις πείσουμε για να απαιτήσουν ε, τα δικαιώματά τους. Τα δικαιώματα υπάρχουν στα χαρτιά αλλά στα χωράφια δεν έχουν δυνατότητα να τα απαιτήσουν. Πώς λοιπόν θα βοηθήσουμε οι μεν γυναίκες, οι γυναίκες ε, νομοθέτηδες, νομοθέτες, πώς θα βοηθήσουμε τις άλλες. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η κυρία Βικτόρια Σμιλούτα Νίλσεν από τη Λιθουανία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και κυρία Τεμπλόβα για την ε, επισκόπηση των στοιχείων του ΩΣΑ που είναι πάντα πολύ ενημερωτικά. Είμαι βουλευτής από την Λιθουανία. Βλέποντας την κατάσταση στη Λιθουανία, από τη μια μεριά έχουμε ένα καλό νομοθετικό πλαίσιο, το νόμο ίσων ευκαιριών και ισότητας. Και επίσης ε, τα ποσοστά απασχόληση μεταξύ ανθρώπων και γυναικών είναι περίπου ταυτόσιμα, οπότε είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό το θέμα. Όμως ε, υπάρχει πολύ ισχυρός διαχωρισμός ε, των επαγγελμάτων για παράδειγμα, οι άντρες ε, στην ε, εκπαίδευση διαλέγουν τα παραδοσιακά ανδρικά ε, πώς το τα παραδοσιακά ανδρικά θέματα εκπαίδευσης, τομείς εκπαίδευσης, ενώ οι γυναίκες κυρίως είναι στα επαγγέλματα τα διδασκαλικά και οι άνδρες κυρίως σε επαγγέλματα επιστήμης και τεχνολογίας και κυρίως υπάρχουν και μερικές ε, προκαταλήψεις που εκφράζονται και στα μέσα για το ρόλο ανδρών και γυναικών. Ποιε χώρες έχουν τη μεγαλύτερη επιτυχία για να λύσουν τα θέματα και του ποσοστού απασχόλησης και των ε, διαχωρισμών των ε, επαγγελμάτων. Πώς θα βοηθήσουμε τις γυναίκες να ασχοληθούν και με τα παραδοσιακά ανδρικά επαγγέλματα και πώς μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό οι βουλευτές. Σας ευχαριστώ από το Μαρόκο. Η κυρία Λομπίνα Έλκολ. Από το Κοινοβούλιο του Μαρόκο. Θα ήθελα καταρχάς να μου επιτρέψετε να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω που είμαστε εδώ σήμερα. Στο Μαρόκο, λοιπόν, έχουν γίνει πολλές μεταρρυθμίσεις όχι μόνο αναφορικά με τις γυναίκες, αλλά και πολλά άλλα ζητήματα που αγγίζουν την κοινωνία. Πολύ ενδιαφέροντα. Και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, την ενσωμάτωση, την ενοποίηση, την ε, ισότητα άντρων και γυναικών. Το τελευταίο σύνταγμα το 2011 έδωσε σημαντική θέση στις γυναίκες. Και πολλά είναι τα νομοθετήματα που αφορούν ακριβώς τις γυναίκες. Τον σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών, την ισότητα των γυναικών. Η κατάσταση είναι ευνοϊκή. Αλλά ασφαλώς πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν και κυρίως ότι αφορά τον οικονομικό κλάδο. Πολλά προβλήματα παραμένουν τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν σταδιακά αλλά και με σαφήνεια για να πετύχουμε τους στόχους μας. Οι γυναίκες λοιπόν στο Μαρόκο περιορίζονται ακόμα σε δραστηριότητε οι οποίες ε, δεν εκτιμούνται ιδιαίτερα στην αγορά εργασία. Οι γυναίκες λοιπόν σε ό,τι αφορά το επίπεδο εκπαίδευσή τους είναι εξαιρετικές. Αλλά έχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η πρόσβαση λοιπόν των γυναικών σε θέσεις ε, ψηλής σημασίας για έλλειψη αποφάσεων είναι προβληματική. Υπάρχει και μια ποσοστό σε ό,τι αφορά τις υψηλοβαθμές θέσεις αυτές, αλλά οι ποσοστώσεις αυτές εξακολουθούν να είναι δύσκολες στην εφαρμογή τους και στην υλοποίησή τους σε τοπικό επίπεδο, στη χώρα μας, σε εθνικό επίπεδο. Και έχουμε επίση ε, ενώσει, συνεταιρισμού γυναικών στο, στην Ήπεθρο. Πάρα πολύ σημαντική εμπειρία αυτή. Πολλέ λοιπόν τέτοιε ε, συνεταιρισμοί. 16% σε επίπεδο εθνικό σε ό,τι αφορά του συνεταιρισμού αυτού. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό σε ό,τι αφορά την Ήπεθρο. Αλλά χρειάζεται ακόμα περαιτέρω προσπάθειε για να υποστρεχθούν αυτές οι γυναίκες οι οποίες ουσιαστικά στηρίζουν οικονομικά τον οικογένειο τους στο σπίτι του και φροντίζουν οικονομικά για όλη την οικογένεια. Πολύ σημαντική λοιπόν η συνταγματική μεταρρύθμιση του 2011, αλλά παραμένουν πολλά τα θέματα τα οποία είναι κρεμή και άλυτα. Σας ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρος. Και τελευταία ομιλήτρια, η κυρία Γιουνές Σιμπή από την Τινησία. Ναι, Λιλιά Γιουνές Σιμπή. Καλημέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι μεταξύ μας για να εορτάσουμε αυτή τη μέρα με πολλές φίλες. Είμαι μέλος του Κοινοβουλίου της Τινησίας και της Επιτροπής Γυναικών. Στην Τινησία η ίση εκπροσώπηση είναι συνταγματικό ε, δικαίωμα. Είμαστε 35% γυναίκες ε, στην, ε, στη Βουλή της χώρας μου, αλλά δεν έχουμε επιτύχει την ισότητα ακόμη. Δεν θα έλεγα ότι τα πάει τόσο καλά η κατάσταση των γυναικών στην Ισία. Το αντίθετο. Ε, από το 2014 προσπαθούμε να πιέσουμε τα Υπουργεία ούτω ώστε οι προπολογισμοί τους να λαμβάνουν υπόψη την διάσταση φύλου. Είμαστε πεπισμένες, οι γυναίκες βουλευτές, καθώς και κάποιοι άνδρες ε, ε, που μας στηρίζουν, είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να γίνει, αλλά δεν καταφέρνουμε να πείσουμε την εκτελεστική εξουσία να το κάνει αυτό. Και το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να τους υποχρεώσουμε. Πώς μπορούμε να τους πείσουμε. Γιατί αν δεν ε, δέχονται την ε, χορήγηση ίσων ευκαιριών στις γυναίκες, αυτό σημαίνει απώλεια για την οικονομία μας που αντιμετωπίζει μεγάλη κρίση. 60% των ε, διπλωματούχων, των πτυχιούχων στη χώρα μου είναι γυναίκες αλλά η κατάσταση εξακολουθεί να είναι άσχημη. Πολλές γυναίκες είναι άνεργοι, είναι άνεργες και παρά το ότι έχουμε πολλούς νόμους που προωθούν την απελευθέρωση των γυναικών, οι γυναίκες ακόμη υποφέρουν, η εργασία, η εργασία τους εξακολουθεί να είναι μη αμοιβόμενη και προσπαθούν να περάσουν αυτούς τους προπολογισμού με βάση και το φύλλο. Ευχαριστώ. Ναι όλες ζούμε σε έναν κόσμο ανδρών εν ολίγης. Θα ήθελα τώρα να ξαναδώσω τον λόγο στην κυρία Τέπλοβα να ολοκληρώσει την συζήτηση και ίσως να δώσει κάποιες απαντήσεις στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ για τις εξαιρετικές αυτές ερωτήσεις και θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι στην δουλειά που κάνει ο ΣΑ ακούμε ε, κάποιες παρόμοιες ανησυχίες ε, ξανά και ξανά να αρχίσω από το τελευταίο σχολείο Πώς μπορούμε να πείσουμε τους ε, κατέχοντες ε, την εξουσία που είναι κατά κανόνα άντρες της χώρας μας ότι η ισότητα είναι μια αξιόλογη επένδυση. Και πάλι λοιπόν επειδή είμαι από τον ΩΣΑ και αυτό που θα σας πω δεν είναι από τη δική μας τη διεύθυνση εμβαθύνουμε ακριβώς ε, στην οικονομική πτυχή και στο οικονομικό επιχείρημα για να δείξουμε ότι ε, το μισθολογικό χάσμα είναι μια χαμένη οικονομική ευκαιρία. Οι γυναίκες είναι ε, ένα μεγάλο σύνολο ανεκμετάλλευτου δυναμικού και Μάλιστα στην Ισλανδία όπου θα γίνει μια διάσκεψη, μια πρόκληση που θα αντιμετωπίσουμε θα είναι ακριβώς ε, και η πλευρά και οι πολιτικοί που ασχολούνται με τον προϋπολογισμό να δουν ε, το θέμα από την σκοπιά του προϋπολογισμού. για το ζήτημα τώρα της ενδυνάμωσης ε, των γυναικών ε, και την δυνατότητα να καταλαμβάνουν αιρετά αξιώματα. Και αυτό το έχουμε αναφέρει και στη δουλειά που κάνουμε και στο Μαρόκο και την Τινησία και σε άλλες αραβικές χώρες και σε άλλες χώρες γενικότερα. Βλέπουμε ότι οπωσδήποτε το ζήτημα είναι πολυδιάστατο. Από την πλευρά της προσφοράς ε, μιλάμε για την αυτοπεποίθηση των γυναικών, τις ικανότητες των γυναικών, την πρόσβαση στα δίκτυα και από την πλευρά της ζήτησης είναι το θέμα του εκλογικού πλαισίου, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση που είναι ένα μεγάλο ζήτημα επίσης και η πρόσβαση στις κοινωνικές υποδομές, γιατί αν δεν υπάρχουν κοινωνικές υποδομές είναι πολύ δύσκολο μετά για τις γυναίκες να κινητοποιηθούν και να αποφασίσουν να κατέβουν υποψήφιες για δημόσια αξιώματα. Και έρχομαι έτσι στην ε, σημασία της ε, ενσωμάτωσης της διάστασης ε, του φύλου στους άλλους τομείς της πολιτικής. Αυτό το οποίο είπα λοιπόν πριν είναι ότι είναι ένας συνδυασμός κατανομής πόρων έτσι όπως δηλαδή δομείται το σύστημα κινήτρων για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα πολιτικά κόμματα, για τις κοινωνικές πολιτικές ε, έτσι θα έλεγα ότι καθορίζεται η υφή της ισότητας. Οπότε αποτελεσματικά εργαλεία ανάλυσης και δεδομένα χρειαζόμαστε σε όλους αυτούς τους ε, τομείς. Γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι πολλές χώρες και ευρωπαϊκές χώρες εστιάζουν ε, στην συλλογή δεδομένων κυρίως τομείς οι, οποίες, οι οποίοι παραδοσιακά συνδέονται με κάποιες με κάποια διάσταση συμμετοχή των γυναικών. Είτε μιλάμε για κοινωνικές πολιτικές, εκπαίδευση, υγεία, αλλά λιγότερα δεδομένα συλλέγονται για τον αντίκτυπο της οικονομικής πολιτική ε, σε άνδρες και γυναίκες, για τις ε, αναδιανεμητικές πολιτικές, ε, τις πολιτικές στέγασης. Τέτοια δεδομένα χρειαζόμαστε για να έχουμε πραγματικά τα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τον αντίκτυπο που έχει η χάραξη πολιτικής. Για τις ε, βέλτιστες ε, πρακτικές, ε, δεν τα λέω με τη σειρά, αυτή τη στιγμή εξετάζουμε τις έρευνες το έχουν κυκλοφορήσει στις χώρες του ΩΣΑ και συλλέγουμε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές που θα είναι διαθέσιμες ε, ως μια εργαλειοθήκη του χρόνου και θα είναι στην σελίδα του όσα σε μια βάση δεδομένων στο διαδικτύο. Για την απλήρωτη εργασία οπωσδήποτε μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν ε, τα μέλη μας ε, σήμερα και γενικότερα θα έλεγα και κάποια από τα εργαλεία, επιλογές που έχουν οι χώρες δυστυχώς ε, δεν είναι νομοθετικά. Μιλάμε για εξτρατείες ενημέρωσης ε, για τον ρόλο της ευαισθητοποίησης, ε, της εκπαίδευσης, να ξεκινάμε από τα νηπιαγωγεία για να ανατρέψουμε αυτά τα στερεότυπα για τους παραδοσιακούς ρόλους ανδρών και γυναικών. Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Ο ρόλος των ΜΜΕ επίσης έχει μεγάλη σημασία και ο ΣΑ κάνει πολλή δουλειά όσον αφορά ακριβώς ε, το πώς οι συμπεριφορές επηρεάζουν την χάραξη πολιτικής και θα δούμε πώς μπορούμε αυτή την ε, πολιτική της ε, παρακίνησης ε, θα λέγαμε μπορούμε να την προωθήσουμε για να αλλάξουν συμπεριφορά και τα νοικοκυριά και να προωθήσουμε την ισότητα για τον διαχωρισμό των φύλων Εκεί όπου βλέπουμε τη μεγαλύτερη βελτίωση είναι στις χώρες όπου υπήρχε η δυνατότητα να επενδύσουν ε, ε, στο να μην υπάρχει χωριστή εκπαίδευση. μεγάλη πρόκληση μεταξύ των μελών του ΟΣΑ είναι η συμμετοχή των ε, κοριτσιών ε, στους, ε, στις θετικές επιστήμες. Και υπάρχουν κάποιες χώρες όπως η Αυστραλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Νέα Ζηλανδία που έχουν κάποιες πρωτοβουλίες για να προωθήσουν την πρόσβαση και την ελκυστικότητα των κλάδων αυτών για τα κορίτσια και βλέπουμε ακριβώς ότι οι διαφορές ε, στις ε, επιλογές εκεί είναι μικρότερες και όπου είναι μικρότερες οι διαφορές είναι μικρότερος και ο διαχωρισμός ε, στον κόσμο της εργασίας κάτι το οποίο μειώνει το χάσμα την ψαλίδα στις πληρωμές. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Νομίζω ότι έχω καλύψει τα περισσότερα στοιχεία. Δύο λόγια για τις ε, ποσοστώσεις. Ε, είναι μια δύσκολη συζήτηση. Το ξέρω και εδώ και στις χώρες σας και γενικά στις χώρες μέλη του ΩΣΑ. Στην ε, σύσταση που ενέκρινε το Συμβούλιο του ΩΣΑ θεωρούμε τις ποσοστώσεις ως ένα από τα μέτρα που μπορούν να λάβουν οι χώρες. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι τρόποι να κλείσει η ψαλίδα, π.χ. υποχρεώσεις ε, δημοσιότητας, ε, εθελοντικές ποσοστώσεις και στόχοι, αλλά ξέρουμε ότι οι ποσοστώσεις ε, έχουν αποτέλεσμα. Οι χώρες οι οποίες έχουν υποχρεωτικές ποσοστώσεις βλέπουν σημαντικές αυξήσεις στις περισσότερες περιπτώσεις. Βεβαίως ε, δεν είναι οι ποσοστώσεις ε, πανάκια, πρέπει να υπάρχουν και μηχανισμοί λογοδοσίας ε, και κάποια κατεύθυνση, ένας προσανατολισμός και εμείς βεβαίως ευχαρίστως βοηθάμε τα μέλη μας με διάφορα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη πρόκληση της ισότητας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να θέσω το θέμα αυτό των ποσοστώσεων. Να πω τι είχε πει ο πρώην Επιτροπός μου. Αρέ... Δεν μου αρέσουν οι ποσοστώσεις, αλλά μου αρέσουν το αποτέλεσμά του το αυτό που κάνουν. Έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι. Και να πω και δύο λόγια μόνο για του τομείς όπου οι γυναίκες εργάζονται, αλλά δεν γνωρίζονται σε εργασία αυτό. Τι βλέπουμε. Και αυτό έχει να κάνει και με τα ποσοστά των γυναικών δικαστών σε όλα τα επίπεδα. Εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση μεγαλύτερη εκπροσώπησης των γυναικών στους τομείς αυτούς. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι. Πέφτουν οι μισθοί, πέφτουν και οι υπηρεσίες και πέφτει και το κοινωνικό κύρος. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να κατανοήσουμε τι συνέπειες έχει η, η, η ισότητα των φύλων και από την άλλη πλευρά. Γιατί όχι μόνο δεν πετυχαίνουμε τον στόχο που επιθυμούμε, αλλά και τελικά α, υπάρχει αντίθετη ε, επίδραση. Δηλαδή, αυτό ισχύει και με τους δασκάλους. Δεν έχουμε τόσο πολλούς άντρες δασκάλους που τελικά θέλετε παρακατιανό επάγγελμα σχεδόν να είναι δάσκαλος κανείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Τέπλοβα, για την εμπειρογνωμοσύνη σας ήταν σαφές ε, είναι σαφή, σαφές ότι έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση, αλλά ακόμα που έχει προσάγκασα από να θεωρηθεί ιδανική. Και θα πρέπει να προωθήσουμε την ισότητα των φίλων περαιτέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. And uh, to the Και προς όλου ε, όλους όσους συμμετείχαν και όλες όσους συμμετείχαν, να σας υπενθυμίσω πρακτικά το εξή. Όσοι θέλετε να πάτε και να παρακολουθήσετε το εργαστήριο υπαριθμών 4, για το κατά πόσο θα υπάρξει ισότητα στην ε, επαγγέλματα μεταξύ ανδρών και γυναικών μπορούν να μείνουν στην αίθουσα. Όσοι θέλουν να πάνε στο εργαστήριο υπαριθμών 5 για την παγκόσμια προοπτική και την ενδυνάμωση των γενικών και οι στόχοι του ΟΗΕ θα πρέπει να πάτε στην προηγούμενη αίθουσα, Γιάν 2Q2. Και θα σας βοηθήσει ένα μέλος από τη γραμματεία της Επιτροπής για την Ισότητα των Γυναικών για να μην χαθείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, πρόσοχή σας, για τη συμμετοχή σας. Σας εύχομαι λοιπόν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση την υπόλοιπη μέρα.